Δείτε ότι εγκρίνονται και αυτές οι αλλαγές. Έχετε λάβει το σχέδιο ημερήσιας διάταξη όπως εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων στις 14 Ιανουαρίου 2010 συμφώνως προς το άρθρο 147 του κανονισμού. Και τώρα θα εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Για την Δευτέρα έχετε κάποια παρατήρηση. Όχι. Οπότε εγκρίνεται η τρίτη για την ε, ημερήσια διάταξη της τρίτης. Επίσης για τα πρόσφατα γεγονότα στην ΑΕΤ προτείνω την εξής αλλαγή αφού συμβουλεύτηκα και τις διάφορες ομάδες. Η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα φύγει από την Τετάρτη το πρωί και θα πάει ως πρώτο σημείο την Τρίτη το πρωί και θα έχουμε επίσης την δήλωση του υπάτου εκπροσώπου και ε, αντιπρόεδρου της Κομισιόν η οποία θα πάει στην θέση αυτή. Ταυτόχρονα από την Τρίτη στην Πέμπτη θα μεταφερθεί η δήλωση του υπάτου εκπροσώπου της, ε, υπάτου του, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δήλωση λοιπόν για τις ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την, Ισία και θα έχουμε δήλωση της Επιτροπής. Οπότε αλλάζουμε απλά τον χρόνο των δύο αυτών σημείων. Η IT πάει στην Τρίτη και η την την Πέμπτη. Παρατηρήσεις? Όχι. Ο κύριος Φόποντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς σας ευχόμαστε καλό έτος. Θα επανέλθετε στο ψήφισμα της ΑΕΤΙΣ γιατί ε, ε, έχει προταθεί ένα ψήφισμα το οποίο νομίζω θα πρέπει να ψηφίσουμε τον Φεβρουάριο. Πράγματι θα το δούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Λοιπόν, δεν έχουμε παρατηρήσει, οπότε μετακινείται η ΑΕΤ στην Τρίτη και η Τινησία θα συζητηθεί την Πέμπτη. Τώρα, όσον αφορά την ε, συζήτηση